για δάνεια σε ξένα ε, νομίσματα. Ο λόγος στον Επίτροπο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τζόναθαν Χίλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα των δανείων σε ξένα χρήματα, σε ξένα νομίσματα. Το να κάνει κανεί ένα στεγαστικό δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι είναι η πιο μεγάλη χρηματοπιστωτική ε, δοσοληψία που κάνουν οι περισσότεροι από εμά στη ζωή μα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ζωντανή και ανταγωνιστική αγορά στεγαστικών δανείων όπου υπάρχουν δυνατότητες επιλογής αλλά όπου ξέρουν και οι καταναλωτές τι παίρνουν και τι κινδύνους αναλαμβάνουν. Ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα, τα δάνεια σε ξένα νομίσματα. Για πολλά χρόνια έχουν δώσει στους καταναλωτές πολύ χαμηλά επιτόκια. Αλλά η πρόσφατη εμπειρία έχει καταδείξει ότι μπορούν να αποτελέσουν και πρόβλημα. Εάν τα δάνεια αυτά τα παίρνουν νοικοκυριά που δεν μπορούν να προστατευτούν έναντι αλλαγών στις ισοτιμίες, στις νομισματικές ισοτιμίες. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα ήταν ένα παράδειγμα. Ήταν πολύ δημοφιλή σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Πολωνία. Όταν όμως η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας σταμάτησε να συνδέει το ελβετικό φράγκο με το ευρώ πέρσι τον Ιανουάριο, το κόστος εξυπηρέτησης αυτών των χρεών ανέβηκε ιδιαίτερα. Και αυτό οδήγησε σε πολλά προβλήματα στα νοικοκυριά τα οποία πρέπει να πληρώσουν να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά του δάνεια και αυτό <clears throat> οδήγησε και σε πίεση στι κυβερνήσει να αναλάβουν δράση και να βοηθήσουν του πιο αναξιοπαθούντε. Ορισμένε χώρε έχουν ήδη περάσει νομοθεσία για το θέμα αυτό και άλλε το εξετάζουν αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με την δράση της Κομισιόν για το μέλλον, εμείς καταρχήν κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με τα δάνεια σε ξένα νομίσματα ε, τη χάνουν καλύτερη διαχείριση για να υπάρχει καλύτερη προστασία του καταναλωτή στην πράξη σύναψη στεγαστικού δανείου. Αυτό όμω δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των υπαρχόντων δανείων σε ξένα νομίσματα. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με κυβερνήσει που και αυτέ θέλουν να ξέρουν ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Προφανώ υπάρχει ανάγκη να προστατευτούν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Αλλά επίση Πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται είναι συνάδων με την ενία αγορά και δεν είναι δυσανάλογα περιοριστικό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία των ε, ευρωπαϊκών εταιρείων να δραστηριοποιηθούν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σκεφτούμε και τον δυνητικό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να γίνει και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών, εάν εμείς υπονομεύαμε την ασφάλεια δικαίου η Κροατία αποφάσισε να εγκρίνει νομοθεσία που επιτρέπει στους ε, δανεισόμενους να μετατρέψουν τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα, σε δάνεια σε ευρώ με την προηγούμενη ισοτιμία πριν ανέβει το ελβετικό φράγκο. Θέτει σε τους καταναλωτές στην ίδια θέση που θα ήταν αν είχαν διαλέξει το δάνειο σε ευρώ. Αλλά το κόστος της ε, μετατροπής που ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ, από ό,τι καταλαβαίνω, τον θέτει στους όμους των τραπεζών, οι οποίες είχαν τότε εκτιμήσει διαφορετικά την ε, ενέργεια αυτή. Δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με την Κομισιόν και φυσικά η κυβέρνηση Κροατίας δεν είχε την υποχρέωση να το πράξει αυτό. Μετά από την έγκριση αυτού του μέτρου έχουμε ελέγξει αν οι τροπολογίες που έφερε η Κροατία στην, στο νόμο της για τα στεγαστικά δάνεια μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι συμβατή με τους κανόνες της ε, ενίας αγοράς. Μπορώ να σας δώσω μια αρχική ανάλυση. Είναι φανερό καταρχήν ότι το να προστατευτούν οι δανειζόμενοι για να αποφευθεί μια κρίση μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμού στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Κατά τη δική μα άποψη, το να επιτρέψουμε σε αυτού οι οποίοι έχουν στεγαστικά δάνεια να τροποποιήσουν τα δάνεια και να περάσουν από το ελβετικό φράγκο σε, ε, σε ευρώ σε μια τεχνητή ισοτιμία με το κόστος να έρχεται αποκλειστικά στους δανειστές μπορεί με να προστατεύσει αυτούς αλλά δεν προστατεύει αυτούς οι οποίοι έχουν δανείσει τα χρήματα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια λύση η οποία είναι πιο αναλογική, σέβεται τις ε, αρχές της ε, συνδίκης και διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Κροατία. Συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση στην Κροατία αλλά και σε άλλε χώρε οι οποίε αυτή τη στιγμή <clears throat> εξετάζουν τη δυνατότητα νομοθεσία προ την ίδια κατεύθυνση. Κατάμε όλε τι ε, επιλογέ ανοιχτέ αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να ξεκινήσουμε και διαδικασίε επί εναντίον τη Κροατία και άλλων χωρών εάν αυτό είναι απαραίτητο. Είμαστε σε επαφή συνεχώς με την κροατική κυβέρνηση και επίσης και με τις αρμόδιες τράπεζες για να μπορέσουμε να βρούμε μια πιο εξορπημένη προσέγγιση ώστε να υπάρξει καλύτερη και δικαιότερη κατανομή του βάρους προσαρμογής. Υποστηρίζω μια τέτοια προσέγγιση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει σύντομα πρόοδος, αλλιώς θα αναγκαστούμε να κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση η οποία εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία, η οποία συνάδει με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύει τους καταναλωτές αλλά επίσης και τις επενδύσεις και την ενιαία αγορά. Αυτή είναι η λύση που προσπαθεί η Κομισιόν να επιτύχει και αυτό θα θέλαμε να γίνει σε όλα τα κράτη-μέλη όπου το θέμα αυτό είναι ένας λόγος ανησυχιών και προβλημάτων. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Τώρα θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο κύριος Καράς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που δώσατε μια απάντηση στο προφορικό μας ερώτημα. Το θέσαμε το προφορικό αυτό ερώτημα γιατί υπήρξε η διαδικασία νομοθεσίας σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, την Πολωνία και στην Κροατία για να μετατραπούν δάνεια σε ελβετικό φράγκο σε ε, ευρώ. Και πολλές φορές είχαν και αναδρομικό χαρακτήρα αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια δικαίου. Το τελευταίο βήμα που έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή μας έδωσε και μεγάλες ανησυχίες για την αξιοπιστία και τη σταθερότητα του πλαισίου δικαίου και σχετικά με αυτό είπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι αυτές οι ενέργειες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην, στον τραπεζικό τομέα και στην πραγματική οικονομία και υπάρχει και κίνδυνος επιμόλυνσης περαιτέρω από τις εμπλεκόμενες χώρες. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια σύνδεση με το θέμα των, ε, του λαϊκισμού. Οι λαϊκιστές θέλουν να έχουν βραχυπρόθεσμα περισσότερες ψήφους, αλλά δεν τους ενδιαφέρει το κράτος δικαίου. Αλλά το κράτος δικαίου είναι ένα από τα θεμέλια τον οποίο έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα κράτος δικαίου και ένα κράτος αξιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να το προασπίσουμε και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε οι δεξιές παρατάξεις να ανατρέψουν και να θέσουν εκτός παιδιάς την ασφάλεια δικαίου. Για τον λόγο αυτό κύριε Επίτροπε θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας θέσω μερικά πρόσθετα ερωτήματα. Έχετε απαντήσει αλλά όχι πλήρως το αρχικό μας ερώτημα. Για ποιες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει να πληροφορηθεί για τις νομοθετικές αυτές προσπάθειες. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Επίσης, ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα θέσετε σε ισχύ για να κάνετε σαφές ότι οι ενέργειες αυτών των κρατών αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων. Έχουμε μια καθαγιασμένη αρχή στην Ευρώπη, όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και η ασφάλεια δικαίου και αυτό ανατρέπεται από το γεγονός ότι ε, ανατρέπεται από την επιστροφή σε, ένα, σε μια ιστορική συναλλαγματική ισοτιμία και όχι στην τρέχουσα συνολοή ε, ισοτιμία. Η Ευρώπη πρέπει να είναι μια κοινότητα δικαίου και ασφάλειας δικαίου. Και πάλι επανέρχομαι για να πω ότι κάποια τέτοια μέτρα τα οποία έχουν βραχυπρόθεσμο λαϊκιστικό χαρακτήρα δεν μπορούν να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίθετα κινδυνεύουν να υπονομεύσουν το οικοδόμημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Καρά. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών Δημοκρατών για 8,5 λεπτά Ιβάν. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά θα τα χρειαστώ τα 8 λεπτά. Φυσικά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρέπει να προστατεύσουμε τις τράπεζες. Είναι σημαντική η ενιαία αγορά, η προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Επίσης και αυτή είναι σημαντική. Όμως, εδώ μιλάμε για μια εμπορική σύμβαση μεταξύ δύο συμβαλωμένων που θα πρέπει να ε, λάβουν ε, και να επομιστούν και τα ε, κέρδη αλλά και τις ενδεχόμενου τους ενδεχόμενους κινδύνους, τα ρίσκα. Οι τράπεζες χορηγούν το δάνειο, παίρνουν επιτόκια, υπάρχει και η ασφάλιση, αλλά επομιστούν και συγκεκριμένους κινδύνους, κάποια ρίσκα να λαμβάνουν. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές για όλους. Πρέπει να δούμε, είναι εδώ ακόμη αντίκτυπος της κρίσης του 2008 το 2006 έως 2008 που τα επιτόκια ήταν 10-12% και τότε είχα συνάψει πολλοί συμπολίτε μας δάνεια ε, στεγαστικά και ήταν και πολύ υψηλέ οι τιμές των κατοικιών. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται και αυτοί οι άνθρωποι για χρόνια αποπλήρωναν τις δόσεις ε, των δανείων, είχαν δώσει μια προκαταβολή 20-30% και όλα αυτά τα χρόνια κατάφερναν οι τράπεζες να παίρνουν ε, τις δόσεις. Όταν όμως δεν ήταν πλέον δυνατό για τους ε, δανειζόμενους να αποπληρώνουν τα δάνεια, πήραν τα σπίτια οι τράπεζες, αλλά κράτησαν και τα δάνεια. Και αυτό είναι μια πραγματική τραγωδία για χώρες όπως η Κροατία ή η Ρουμανία. Και είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού. Στη βάση της οικονομικής κρίσης του 8 ήταν οι τράπεζες, αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Οι τράπεζες μεταμορφώθηκαν σε επενδυτικές τράπεζες που έδιναν στεγαστικά δάνεια χωρίς καν μία δικλίδα ασφαλείας και έδιναν δάνεια και σε άτομα που ήξεραν ότι δεν πρόκειται ούτε δέκα ζωές να ζούσαν να αποπληρώσουν αυτά τα δάνεια. Αυτή λοιπόν η διάθεση, αυτή η απληστία των τραπεζών είναι αυτή που δημιούργησε το πρόβλημα. Οι διοικητές των τραπεζών και των επενδυτικών τραπεζών κράτησαν τα κέρδη, αλλά άλλοι έχασαν τα σπίτια τους γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις δόσεις που κατάφεραν παρόλα αυτά πριν την κρίση να τις ε, πληρώνουν για δεκαετίες. Και όχι μόνο τους πήραν τα σπίτια, αλλά τους υποχρεώνουν να αποπληρώσουν το δάνειο και από πάνω. Να βάλω αυτή την τιμή του ενός ε, δις ε, και το βάζω εντός αγωγικών που πρέπει να ε, καταβληθεί κατά κάποιο τρόπο για να αναλάβουν και την ευθύνη τους οι τράπεζες και να ρυθμιστεί η κατάσταση. Αλλά υπάρχει... δεν υπάρχει μόνο αυτό το νούμερο. Πρέπει να δείτε και άλλα νούμερα. Και ποιο ήταν το κέρδος των τραπεζών και ποιο ήταν το ύψος των δανείων που χορηγήθηκαν και ποια είναι η αξία ε, του, των ακινήτων ε, τα οποία πήραν από πελάτες τράπεζες και δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν πλέον το δάνειό τους. Και αυτά τα ακίνητα, αυτή η περιουσία, ε, πώς τη χρησιμοποίησαν τράπεζες στην αγορά ακινήτων. Τώρα για τη Ρουμανία συγκεκριμένα υπήρξαν κάποιες τράπεζες που πήραν ε, τα σπίτια αυτών που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το δάνειό τους και τα έδωσαν σε άτομα που τελικά τα πούλησαν για μια δεκάρα και τα πήραν άνθρωποι που είχαν σχέσεις με τις ε, τράπεζες αυτές. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό ως φαινόμενο. Δημιουργεί στρεβλώσεις στην οικονομία, στην αγορά που αναφέρατε και εσείς ο ίδιος. Δεν μιλάμε μόνο εδώ για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, μιλάμε και για την ευθύνη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ε, για την ευθύνη των τραπεζών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι τράπεζες όταν ε, έχουν δώσει κάποια δάνεια. Κανείς δεν απαγορεύσει μια τράπεζα να πάρει περαιτέρω μέτρα ασφαλείας. και μπορεί ο πελάτης επίσης να επιλέγει. Γιατί υπήρξε ένας ε, νόμος πρόσφατα στη Ρουμανία. Ε, τι θα κάνει. Να δώσει περαιτέρω εγγύηση ή να επιστρέψει το σπίτι. Στη Ρουμανία πλέον αν ένας πολίτης δεν μπορεί να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο που έχει συνάψει, μπορεί να επιστρέψει στην τράπεζα το οίκημα αυτό και έτσι να αποπληρώσει το χρέος του κατά κάποιο τρόπο. Αυτό βέβαια ε, δημιουργεί πρόβλημα προβλεψιμότητας για τους επενδυτές και είναι αρνητικό, ναι, αλλά στην Δανειακή Σύμβαση ξεκάθαρα λέγεται ότι η υποθήκη καλύπτει ε, την αξία του δανείου. λοιπόν που επιστρέφεται το διαμέρισμα ή το σπίτι στην τράπεζα πρέπει και να κλείσει η υποθήκη. Λέτε ότι ήταν μεγάλες οι απώλειες για τις τράπεζες. Ποιες ήταν αυτές οι απώλειες, σαν ένα άτομο, ένας άνθρωπος ε, κανονικός, πληρώνει 30% προκαταβολή, πληρώνει τους τόκους και τις δόσεις του κεφαλαίου επί χρόνια, πληρώνει και τη διαφορά της συναλλαγματικής οντιμία, αλλά μετά δεν μπορεί μετά από 2-3 χρόνια να πληρώσει. Έχει πάρει ήδη τις δόσεις τη οι τράπεζες, έχει πάρει την προκαταβολή και παίρνει και το σπίτι. Ποια είναι η απολιά τη λοιπόν, δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ξεκάθαρες αυτές οι συμβάσει, ώστε να μπορούν όλοι να ε, αναλαμβάνουν και τι ευθύνε του και ε, ανάλογα να έχουν και το σχετικό κέρδος. Ευχαριστώ πολύ. για την ομάδα των συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Ο κύριο Τσαμπάσκι έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι ενδιαφέρεστε για την υπόθεση αυτή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ορισμένες χώρες μέλη Πολλοί χρησιμοποίησαν τα ελβετικά φράγκα, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από ότι βγήκε στο τέλος το 60% των μη εξυπηρετούμενων δανείων απεδείχθη ότι ήταν σε ξένο νόμισμα. Περιέργως το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο ε, είναι χώρες που έχουν δώσει δάνεια σε πολίτες άλλων χωρών, γιατί είναι διεθνή χρηματοδοτικά κέντρα βέβαια οι δύο αυτές πόλεις. Έχουν ε, ίσως χαμηλότερα επιτόκια, έχουν ε, μακρά περίοδο απόσβεσης, αλλά δεν πάβει να είναι μια επικερδής δραστηριότητα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φυσικά οι πελάτες τους υφίστανται τους κινδύνους τους συναλλαγματικούς. Το 2008 έπεσε σε σχέση με το ελβετικό φράγκο η αξία πάρα πολλών νομισμάτων και ήδη από τότε πολλοί που είχαν δανειστεί σε ελβετικά φράγκα αναγκάστηκαν να επιστρέφουν κάθε μήνα πολύ περισσότερα χρήματα. Στη Βουλγαρία σαν παράδειγμα Πολλά από τα δάνεια ήταν σε ελβετικά ευρώ, αλλά τον τελευταίο καιρό αυτό έχει αλλάξει και ε, τα δάνεια είναι πλέον τα στεγαστικά τουλάχιστον σε ευρώ ή στο εθνικό βουλγαρικό νόμισμα. Ιδιαίτερα τώρα που το ευρώ έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Νομίζω ότι η νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τις δυνατότητες για να διορθωθούν οι άδικες ρήτρε των δανείων αυτών. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο. Στην κυρία Ματιάς, έξι λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε έχουμε ένα θέμα ενώπιό μας το οποίο για ορισμένους είναι τεχνικό και πολύ ειδικό αλλά μιλάμε για ένα βασικό πρόβλημα ουσίας και πολιτικής το οποίο συνδέεται με πολλά άλλα ζητήματα. Νομίζω ότι καταρχήν η διατύπωση αυτού του, αυτής της συζήτησης είναι λαθασμένη. Έχουμε να κάνουμε με δάνεια τα οποία έχουν γίνει σε εθνικά νομίσματα τις περισσότερες φορές και όχι σε ξένα νομίσματα που οδήγησαν σε προβλήματα. Μία από τις ε, πρακτικές που διακηρύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πρέπει να φύγει κάθε είδος κινδύνου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να περάσει τους ώμους των καταναλωτών και των δανειζομένων. Ο μόνος λόγος για τον οποίο είναι ε, η τραπεζική δραστηριότητα κερδοφόρα είναι γιατί επομίζονται τα τραπεζικά ιδρύματα ένα τμήμα του κινδύνου που υπάρχει πάντα στις χρηματοπιστωτικές δοσοληψίες. Αυτό πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη σε οποιαδήποτε συμφωνία. Σε οποιαδήποτε και συγκεκριμένα για τις στεγαστικές για τη στεγαστική πίστη. Και εδώ έχουμε την περίπτωση ε, χιλιάδων οικογενειών που είναι σε τραγική κατάσταση, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, χρειάστηκε να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και παρόλα αυτά ακόμα πρέπει να ε, πληρώνουν όλα αυτά γιατί είναι απόλυτα προστατευμένος ο πιστοτικός τομέας. Από την άποψη αυτή η απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου για το συγκεκριμένο αυτό θέμα είναι αρκετά εύγλωτη. Είναι εύγλωτη για τη στάση που κατούν οι ευρωπαϊκοί δεσμοί σε σχέση με τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρέμβουν στην λειτουργία των εθνικών χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως έχουν κάνει με παράνομο τρόπο στην περίπτωση πώληση τραπεζών στην Πορτογαλία, για συγκεκριμένες τράπεζες. Αν όμω υπάρξει ένα πολίτη ο οποίο καταγγείλει μια συμφωνία δανείου επειδή δεν τηρεί την ε, ε, αρχή της δικαιοσύνης και της καλής πίστης, η απάντηση της Κομισιόν είναι όχι. Θα πρέπει να πάτε την τράπεζα στα δικαστήρια και να τα βρείτε. Έχουμε λοιπόν αυτή την Ευρώπη, η οποία έχει τιτανική δύναμη για την εφαρμογή λιτότητος και περιορισμού των εθνικών ε, προϋπολογισμών, πάντα προσπαθεί να προστατεύσει τους ε, μεγάλους και όχι τους μικρούς, τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους έναντι των απλών πολιτών. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε, μεταξύ άλλων, είναι και η δημοφιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει καταβαρθρωθεί το τελευταίο καιρό. Καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτούς οι πολίτες και όλα αυτά τα προσχήματα και τις δικαιολογίες που προβάλλουν οι χρηματοπιστωτικοί φορείς θα καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι δεν έχουν καμία αξία. Θα πρέπει να προστατεύσει η Κομισιόν όμως του καταναλωτέ. Θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη δράση της Κομισιόν για να προστατεύσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μονάχα την ελεύθερη αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Δίνω τώρα τον λόγο από τους μη εγγεγραμμένους στην κυρία Κριστίνα Μορβάη. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Περίμενα με ανυπομονησία τη σημερινή συζήτηση και ούτε τα μάτια μου δεν ε, μπορώ να πιστέψω ότι συζητούμε τα στεγαστικά δάνεια και άλλα δάνεια σε ξένο νόμο επιτέλους Ανοίξατε τα μάτια σας οι ευρωκράτες. Βαρεθήκατε τις εκατοντάδες επιστολές διαμαρτυρίας από συμπολίτες μας που φτάσανε στα πρόθερα της αυτοκτονίας επειδή ε, δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο, πολύ απλά. Εδώ στην Ευρώπη πολλές χιλιάδες άνθρωποι ζουν υποκαθεστώς σύγχρονης δουλείας για, δουλεύουν και ζουν για να πληρώνουν τα δάνεια στις τράπεζες. Αυτό ε, αφορά πάρα πολλές οικογένειες στην Ευρώπη. Εσείς εδώ, οι Βρυξέλλες, η Ευρώπη που θέλετε να βάζετε τη μύτη σας παντού και να, και να χώνετε τα χέρια σας παντού. Ξυπνήσατε τώρα. Τι θέλετε όμως τελικά. Αυτό που θέλετε είναι να ξεκινήσετε διαδικασίες επί παραβάση κατά της Κροατίας, για παράδειγμα, διότι πήρε το μέρος των πολιτών ε, το κρατικό κράτος και όχι το μέρος των τραπεζών. Εμείς είμαστε στο πλευρό της Κροατίας, τη στηρίζουμε μέχρι σε σχάτων. Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε κατά τα άλλα. Γιατί έχετε στενές διασυνθέσεις με οικονομικούς εγκληματίες, με το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή μαφία δεν ξέρω πώ κοιτάζεστε στον τραπέζι, στον καθρέφτη, θα έπρεπε να ντρέπεστε και εσεί, κύριε Επίτροπε. Τι θα κάνετε για τον κόσμο. Θέλετε να σώσετε και να στηρίξετε τι τράπεζε, αλλά πώ θα σώσετε και θα στηρίξετε του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Ποσπισίλ, μέχρι πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που προηγήθηκε είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι κρίμα που το συζητάμε πέμπτη απόγευμα. Επίτροπε, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία μας είπατε και είμαι ικανοποιημένος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι σημαντικό να έρθει σε επαφή με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών που προτείνουν ειδικέ ρυθμίσεις σε σχέση με τις συναλλαγματικές αυτές ισοτιμίες. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται κοινωνικά σε δύσκολη κατάσταση, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να βλαθεί και η ενιαία αγορά. Οι λύσεις που θα δοθούν δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον τομέα αυτό. Κατανοώ αυτούς οι οποίοι δανείστηκαν χρήματα σε ξένο νόμισμα. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει ε, στο να υιοθετήσουμε νομοθετικές ρυθμίσεις εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό ε, με ικανοποίηση όπως είπα άκουσα την παρέμβαση του κυρίου Χίλ. Αν κάποιες κυβερνήσεις θέλουν να βοηθήσουν τους πολίτες που διατρέχουν κίνδυνο και πήραν ένα βολικό σε εισαγωγικό δάνειο που τελικά δεν ήταν και τόσο βολικό, δεν θα πρέπει να το κάνουν εις βάρος ε, των επιχειρηματικών ομίλων των διαφόρων χωρών και εις βάρος άλλων ομάδων που έχουν δανειστεί χρήματα. Αν πάρουμε ειδικά μέτρα για αυτούς, τότε οι άλλοι που δεν δανείστηκαν σε ξένο νόμισμα τι θα πούν. Ας μην βοηθήσουμε λοιπόν κάποιους για να θίξουμε τους υπόλοιπους. Εγώ προέρχομαι από την Τσεχία, λέει ο κύριος Ποσιμπίλα. Μιλάμε για την Ανατολική Ευρώπη. Όταν υπήρξε ένα μπούμ σε τέτοια δάνεια, στη χορήγηση τέτοιων δανείων, εγώ ήμουνα μέλος της κυβέρνησης της Τσεχίας και προειδοποιούσαμε τους Τσέχους πολίτες ε, για αυτές τις πολύ ωραίες υποσχέσεις αυτών που πουλάγαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τα πράγματα στην Τσεχία, παρότι είμαστε μικρή χώρα, έχουμε μια ισχυρή οικονομία, έχουμε ισχυρές τράπεζες και λίγα προβλήματα σε σχέση με τους γείτονες γύρω από το θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσον προειδοποίησαν οι χώρες αυτές τους πολίτες ότι παίρνοντας αυτά τα ελκυστικά δάνεια ε, στην ουσία ήταν σε διαδικασία να αυξήσουν τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν οι πολίτες τους. Ας βρούμε λοιπόν λύσεις που δεν θα θίξουν την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο που σεβαστήκατε το χρόνο σας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Σον Κέλλη για τρία λεπτά. Αμάν λάθος έκανα. Κανείς δεν είναι τέλειος λέει ο πρόεδρος, έκανα λάθος και κανονικά τώρα έρχεται η σειρά του κυρίου Μαμίκινς. Έχει οκτώ λεπτά κύριε Μαμίκινς. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δει κανεί ε, την κατανομή των ε, συναλλαγμάτων υπάρχει μια σχέση που έχει να κάνει με το εμπόριο και την χρησιμοποίηση αυτών των ε, νομισμάτων. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν έξω από τα σύνορά του το δολάριο, το ευρώ, το γεν, το αυστραλιανό δολάριο, το ελβετικό φράγκο, την αγγλική λίρα κτλ. Το ίδιο έχει να κάνει και με την δανειοδότηση βάσει της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιανουάριο του 2016 τα περισσότερα δάνεια σε ξένο νόμισμα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε δολάρια και ελβετικά φράγκα. Τα, τα νοικοκυριά είναι σημαντικοί δανειστές μετά από τους χρηματοπιστωτικούς τορί Σε πολλές χώρες μπορούν να κάνουν δάνεια ε, σε άλλα νομίσματα και στην περίπτωση της Πολωνίας αυτό είναι η πλειοψηφία. Σε άλλες χώρες όμως όπως είναι η Τσεχική Δημοκρατία και η Πολωνία δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου δάνεια σε ξένο νόμισμα ενώ σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο και η Κύπρος το μεγαλύτερο μέρος των δανείων γίνεται από χρηματοπιστωτικούς τομείς. Στην Πολωνία και την Ελλάδα τα μισά περίπου δάνεια είναι σε ξένο νόμισμα, με άλλα λόγια. Εξαρτάται από την κατάσταση οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοπιστικής σταθερότητας και άλλους παράγοντες, το ποια επιλογή θα διαλέξουν οι καταναλωτές <clears throat> για να δανειοδοτηθούν. Στην περίπτωση λοιπόν που υπάρχει ένα δάνειο σε άλλο νόμισμα, με σταθερούς όρους αποπληρωμής, με ε, υπάρχει μια, μπορεί να υπάρχει μια προαίρεση για ανταλλαγή των δύο νομισμάτων σε σταθερή ισοτιμία. Αλλά δεν καλύπτει αυτό όλα τα δάνεια αυτού του είδους και αυτή είναι και η πηγή του προβλήματος και γι' αυτό χρειάζεται ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό σύστημα για να δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου οι δανειστές γνωρίζουν πλήρως τους κινδύνους τους οποίους ε, επομίζονται ενώ οι τράπεζες φυσικά δεν μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού. <clears throat> Ο κύριος κίνδυνος σε περίπτωση δανείου σε ξένο νόμισμα είναι ο κίνδυνος ο οποίος έχει να κάνει με την πτητικότητα, με, την, το ευμετάβλητο των ε, συναλλαγματικών ισοτιμιών. Παραδείγματος χάρη η ιδανική κορώνα είναι συνδεδεμένη με το ευρώ. Αλλά αν έχουμε ένα άλλο νόμισμα το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με το ευρώ, ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κανείς να ασχολείται και με το θέμα αυτό. Αν πάρει κανείς ένα δάνειο <clears throat> παραγωγικά στην Ουκρανία ή στην ε, Ρωσία σε δολάρια ή σε ευρώ πριν από μερικά χρόνια, αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές λόγω ακριβώς της ε, υποτίμησης του ουκρανικού και ρωσικού νομίσματος τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να προκύψουν σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση ξένων νομισμάτων όταν υπάρξει μια χρηματοπιστωτική κρίση ή μια οικονομική κρίση σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου εξετάστηκε το θέμα της επιστροφής στη δραχμή από τους φορείς τους χρηματοπιστωτικούς. Σε περιπτώσεις όμως που γίνεται μια, μια δανειοδότηση σε σταθερό σε σταθερή ισοτιμία σε σχέση με το εθνικό νόμισμα, τα προβλήματα αυτά έχουν ε, ελαχιστοποιηθεί. Πρόσφατα ετέθη ένα ερώτημα προς την Κομισιόν για το θέμα των ε, δανείων αυτών σε ξένα νόμισμα ή καλύτερα των αναδρομικών προσαρμογών δανείων σε ξένα νομίσματα στο εθνικό νόμισμα. Αυτό αφορούσε χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές οι πολίτες εκεί πήραν δάνεια προσωπικά τα οποία είναι σε ξένο νόμισμα και με τον τρόπο αυτό πολλά νοικοκυριά βρέθηκαν σε κίνδυνο να αντιμετωπίσουν προβλήματα εάν υπήρξε ταχεία μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πάρα πολλοί επίσης είχαν και στεγαστικά δάνεια σε ξένα νομίσματα. Για αυτό το λόγο μπορεί να είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η εθνική χρηματοπιστωτική σταθερότητα η οποία κινδυνεύει από τέτοιες ενέργειες. Ένας από τους με τον οποίο έγινε αυτό είναι να επιβάλλουν τα κράτη, να δώσουν μάλλον τα κράτη δυνατότητα να υπάρξουν αναδρομικές <clears throat> προσαρμογές με παλιές συναλλαγματικές ε, ισοτιμίες. Αυτό όμως θέτει το θέμα της συμμόρφωσης με την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ελευθερία εγκατάσταση και ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Γιατί υποσκάπτεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εσωτερική αγορά. Επομένως, ε, πρέπει να επισημάνω ότι δεν καλύπτονται ακόμα τα θέματα αυτά από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον όμως η Κομισιόν είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θα είναι απαραίτητο η Κομισιόν να κάνει σαφή τη θέση της για το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τη νομική συμβατότητα της πρακτικής αναδρομικής ε, ανταλλαγής δανείων σε ξένο νόμισμα με δάνεια σε εθνικό νόμισμα σε ιστορικές ισοτιμίες και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, θα έπρεπε να αναφέρω ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο θα είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια νομοθετική κάλυψη σε όλες τις συμφωνίες δανείων που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαμίκη. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Στάνισλαβ Πόλτσακ, έχει το λόγο για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά λυπάμαι και το παραλαμβάνω λυπάμαι που συζητούμε ένα τόσο σημαντικό θέμα ε, μια πέμπτη απόγευμα. Βέβαια από την άλλη με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσα όσα είχε να μας πει ο Επίτροπος με βάση τις δηλώσεις του είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά το θέμα και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερος. Παρότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι πολλά ακόμη μπορούν και πρέπει να γίνουν. Αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα στην τσεχική δημοκρατία ε, δεν είναι τόσο σοβαρό ίσως, αλλά πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης και όχι μόνο, ε, πλήγησαν πολύ σκληρά από αυτό το πρόβλημα. Ήταν πολύ ενδιαφερόμενοι ε, για αυτά τα δάνεια σε ξένο και πολλές φορές τελικά, ε, επειδή ήταν πολύ χαμηλά τα επιτόκια, τα προτίμησαν και τελικά κατάληξαν αυτοί που γνωρίζουμε λόγω των διακυμάνσεων, ε, και μπορεί και να μην άλλαξε τελικά ε, το επιτόκιο. Χρειάστηκε να πληρώσουν ε, παρόλα αυτά οι δανειζόμενοι πολύ μεγαλύτερα ποσά και σε κάποια κράτη με, λόγω αυτού του προβλήματος και του μεγέθους που είχε αποφάσισαν να λάβουν κάποια μέτρα αναδρομικά και τα μετέτρεψαν σε δάνεια σε τοπικό νόμισμα αυτά τα δάνεια σε ξένο Και τώρα βλέπουμε ότι υπονομεύεται κατά αυτόν τον τρόπο μία από τι βασικέ ε, αξίε και αρχέ τη Ένωση που είναι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Και επίση ε, δεν γίνεται, βλέπουμε να μην τηρείται το κράτος δικαίου. Αυτά τα κατανοώ. Κατανοώ επίσης γιατί επέλεξαν τα κράτη-μέλη αυτόν τον τρόπο για να επιλύσουν αυτές τις πολύ λεπτές ε, καταστάσεις. Όμως ε, η αναδρομική ισχύς αυτών των μέτρων θα πρέπει να καταδικαστεί. Θα πρέπει η πρόληψη να υπερτερεί της θεραπείας. Και θα πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ε, δανειζομένων και όχι να λαμβάνονται δραστικά μέτρα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ούτε βέβαια και να υπονομεύσουν ε, την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Φυσικά και γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα προβλήματα, όπως είναι η κατάχρηση ορισμένων άρθρων των ε, δανειακών συμβάσεων. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται διαφορετικά επιτόκια Μάλιστα και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιλήφθηκε ορισμένων υποθέσεων και με τις αποφάσεις που έλαβε ακυρώθηκαν κάποιες από αυτές ε, τις συμβάσεις που ήταν ε, εποφελείς μόνο για τις τράπεζες. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Χαίρομαι κύριε Επιτροπή γιατί θεωρώ ότι πράγματι πρέπει να αναγνωρίσουμε και να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών χωρίς όμως να υπονομεύσουμε τις αρχές του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ. Σον Κέλλη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ικανοποιημένος ιδιαίτερα που μπορώ να μιλήσω για το θέμα αυτό εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας. Όταν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται ιδιαίτερα χαμηλά, πιο χαμηλά από ποτέ, Βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, τα επιτόκια τα οποία χρεώνουν ε, οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα ψηλά. Στην Ιρλανδία 4% χρεώνουν ε, οι τράπεζες ενώ ο μέσος όρος σε άλλες χώρες είναι γύρω στα 2,5%. Αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε θέσει και στον Τράγκη και περιμένουμε την απάντησή του. Η συζήτηση σήμερα όμως μου δημιουργεί και περισσότερες ανησυχίες. Πολλοί Ιρλανδοί θεωρούν ότι τα δάνεια σε ξένο νόμισμα σημαίνει χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερη περίοδος ε, ε, επιστροφής, αποπληρωμής. Αυτό όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ προσεκτικά Υπάρχουν κίνδυνοι στην διαδρομή και οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε αποπλερωμές πολύ μεγαλύτερων ποσών. Πρέπει λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές, δανειολήπτες να είναι σίγουροι και σωστά ενημερωμένοι. Ξέρουμε ότι όταν τα δάνεια είναι σε ξένο νόμισμα και όσο περισσότερα είναι αυτά η οικονομία γίνεται ασταθέστερη και αυτό επηρεάζει και την κατανάλωση και τη ζήτηση στον τομέα της κατοικίας. Και γι' αυτό περισσότερες τέτοιες μορφές δανειοδότησης θα δημιουργήσουν περισσότερη αστάθεια γιατί επηρεάζονται από μια ιδιαίτερα πτητική ισορροπία στις ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάρα πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια με ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό. Και τώρα που οδηγούνται οι Βρετανοί προς το Brexit, εάν υπάρξει κάτι τέτοιο, οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να δημιουργήσουν νέες ρυθμίσεις για να κρατήσουν σταθερή την οικονομία τους ε, σε μια δύσκολη περίοδο. Γι' αυτό ακριβώς η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπεύθυνη στάση των συμβαλωμένων σε δανειοληπτικές δραστηριότητες είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμο ιδιαίτερα από την πρόσφατη ιστορία. Να πω προς τον κύριο Επίτροπο ότι η δουλειά την οποία κάνει είναι καλή δουλειά και του ευχόμαστε συνέχεια και σταθερότητα στην προσπάθειά του η οδηγία για τα δάνεια πρέπει να προσέχετε γιατί πραγματικά πολλές φορές είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά αλλά απίσω από αυτό κρύβονται πολλοί κίνδυνοι. Ευχαριστώ, πολύ πολύ Πρόεδρος.